ότι η Επιτροπή ε, παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς ε, την κατάσταση και προτίθεται να βοηθήσει και την Ιταλία και την Τινησία και τις άλλες χώρες όπως προκύπτει. Ευχαριστούμε κυρία Μάλστρομ και με την παρέμβασή σας ολοκληρώνουμε τη συζήτηση αυτή και τώρα στην ημερήσια διάταξη περάμε στην έκθεση της κυρίας ε, Όμεν Χόιτεν πάλι στα θέματα των επαρκών, βιώσιμων και ασφαλών ευρωπαϊκών ταξιδιωτικών συστημάτων στην Ευρώπη. Δίνω λίγο χρόνο για να αλλάξουν θέσεις οι επίτροποι Ψάχνουμε την κυρία εισηγήτρια. Πολύ ωραία. Θέλω να δώσω λοιπόν το λόγο στην εισηγήτρια για να το παρουσιάσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για την ευχάριστη και επικοδομητική συνεργασία και βεβαίως και τη γραμματεία του Κοινοβουλίου και τους δικούς μας συνεργάτες. Δεν ήταν απλό αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Υπήρχαν πάρα πολλές τροπολογίες και θεωρώ πως τα καταφέραμε γιατί τώρα έχουμε μια καθαρή αντίδραση στην πράσινη βίβλο. Για να έχουμε λοιπόν επαρκή βιώσιμα και ε, ασφαλή ευρωπαϊκά συνταξιωτικά στήματα όπως θέλει ο Ευρωπαίος πολίτης. Αυτό δεν είναι κάτι το απλό και εξακολουθεί να παραμένει ευθύνη των κρατών μελών. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν επιτρέπεται να κάνουμε προτάσεις μέσω της μεθόδου του ανοιχτού συντονισμού. Κυρία Πρόεδρε, η βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών στήματων είναι υποπίεση. Έχουμε μια αντίστροφη ηλικιακή πυραμίδα. Έχουμε περισσότερους ηλικιωμένου που ζουν περισσότερο και μικρότερο ρυθμό εργαζομένων. Τα συστήματα του πρώτου πυλώνα είναι τέλεια έκφραση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών και θα παραμείνουν σημαντικό κομμάτι και στο μέλλον. Αλλά το βάρος για τις νέες γενιές είναι πάρα πολύ μεγάλο και ασκεί πίεση στους συλλογικούς προϋπολογισμούς και αυτό βεβαίως αντικατοπτρίζεται και στο Σύμφωνο Σταθερότητας είτε το θέλουμε είτε όχι. Κυρία Πρόεδρε, τα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης. Προτάσεις οι οποίες υπήρχαν για να καταλήξουμε σε μια ευρωπαϊκή σύνδεση των ε, ορίων αυτών με το προσδόκιμο ζωής, τις απορρίπτω. Και αυτό το απορρίπτω γιατί διαφέρει το προσδόκιμο ζωής στα κράτη-μέλη. Και αν είναι να κάνουμε κάτι τέτοιο, νομίζω πως δεν θα είναι και πάρα πολύ κοινωνικό. Αυτό το οποίο θεωρούμε είναι πως θα πρέπει να πάμε βέβαια προς μια λογική ηλικία συνδεξιοδότησης, αλλά αυτό θα γίνει από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους και σε επίπεδο κράτους μέλους. Επίσης υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, κυρία Πρόεδρε, δηλαδή το ότι θα πρέπει να φροντίσουμε να παραμείνουν οι ηλικιωμένοι στη δουλειά και να υπάρχουν έτσι πιο ευέλικτες σταδιοδρομίες και πιο ευέλικτοι κανόνες για την σύνταξη και να μπορέσουμε να προσαρμόσουμε βέβαια και τις συνθήκες για να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται οι ηλικιωμένοι. Υπάρχει βεβαίω και ο δεύτερο πυλώνα, ο οποίο έχει κάνει πάρα πολλέ οικονομίε. Γιατί ξέρετε, ορισμένε φορέ αυτό γίνεται από κοινού μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, άλλε φορέ από τα κράτη-μέλη. Υπάρχουν λοιπόν τα ε, συστήματα αυτά τα οποία εξοικονομούν για το μέλλον και βεβαίως ε, είναι σε καλύτερη, σήμαση, σε καλύτερη μοίρα από τα δημόσια συνταξιδοτικά συστήματα. Όμως και εκεί πέρα ε, ασκεί πίεση ο ηλικιωμένος πληθυσμός. Οπότε βλέπετε πως υπάρχουν εδώ πέρα κάποιες εγγυήσεις οι οποίες ε, αφορούν τις μελλοντικέ συντάξεις. Οπότε θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρότερες απαιτήσει φερεγγιότητας. Οι τωρινέ δεν είναι επαρκείς. Πρέπει να υπάρχει καλύτερη υποπτία, καλύτερη λειτουργία του συστήματος, αλλά πρώτα απ' όλα μια σωστή και εις βάθος ανάλυση της φερεγγιότητας των συνταξιδοτικών αυτών ταμείων. Δεν θα περάσουμε τώρα στην συζήτηση ε, για τα παράγωγα. Δεν μπορούν να συνδεθούν τα παράγωγα με τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Δεν είναι εκεί πέρα για κερδοσκοπία τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Ο τρίτος πυλώνας τώρα, κυρία Πρόεδρε, δεν πρέπει να έχουμε πάρα πολύ μεγάλες προσδοκίες. Αυτές ε, τις δυνατότητες αποταμίευσης μπορεί να τις εκμεταλλευτεί κανείς αν έχει λεφτά, αλλά θέλουμε να δημιουργήσουμε περισσότερη συνείδηση στον κόσμο, ενημέρωση του κόσμου για τη σύνταξή του. Οπότε πρέπει να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά τον τρίτο πυλώνα και την ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά. Κατόπιν, για την επάρκεια. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρέπει να το δουν τα ε, κράτη-μέλη. Κατόπιν, διασυνοριακή λειτουργικότητα. Βλέπετε πώς θα πρέπει να μην βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση οι εργαζόμενοι εκείνοι οι οποίοι κινούνται από χώρα σε χώρα. Αυτά και όπως σας είπα θα πρέπει να κάνουμε μια μελέτη για τις επιπτώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ να είστε πολύ προσεκτικοί με το λόγο γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Λοιπόν, ο κύριος Επίτροπος, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, κυρία Συγήτρια. Η πράσινη βίβλος για της συντάξης που εκδόθηκε πέρσι το καλοκαίρι ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση και απαραίτητη συζήτηση για τις συντάξει στην Ευρώπη. Κάνουμε πάνω από 100 συναντήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη και λάβαμε περίπου 1.800 απαντήσεις στα όσα έχουμε στην ανακοίνωση αυτή η οποία περιγράφει τις βασικές προκλήσεις και διατυπώνει 14 ερωτήματα για το πώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε να είναι ασφαλείς, επαρκείς και βιώσιμες οι συντάξεις. Βεβαίως πάντοτε σεβόμενοι την αρχή της επικουρικότητας. Ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην Πράσινη Βίβλο γιατί οι Επίτροπη Ρεν Μπαρνιέ αλλά και εγώ ίδιος θεωρούμε πως τέτοιου είδους συντάξεις χρειάζεται συντονισμένη δράση ε, και συντονισμένες πολιτικές σε τρεις ε, κυρίως ε, χώρους ευθύνης. Και θα ήθελα να σας αναφερθώ στα όσα εκδώσαμε πέρσι. Καταρχήν πρέπει να ξεπεράσουμε αυτή την έλλειψη ισορροπίας που υπάρχει μεταξύ προσδόκιμου ζωής και ηλικία συνταξιοδότησης. Δεύτερον, θα πρέπει να προσαρμόσουμε ε, την τακτική μας γιατί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις μεταρρυθμίσεις των συνταξιδοτικών συστημάτων που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία 10 χρόνια στην Ευρώπη. Και τρίτον, χρηματοπιστωτική κρίση. Είδαμε τι σημαίνει έκθεση στις αγορές και θα πρέπει να έχουμε συνταξιοδοτικά σύστηματα τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη την εξασφάλιση έναντι κινδύνων και θα δίνουν τη δυνατότητα απορρόφησης ε, σοκ και κρίσεων. Θέλουμε συστήματα τα οποία θα λάβουν υπόψη και την επιταχυνόμενη γύρανση του πληθυσμού. Τα κράτη-μέλη ήδη αυτή τη στιγμή συνεργάζονται μεταξύ τους εδώ και καιρό για να ανταλλάξουν εμπειρίες και βέλτιστες πρακτικές στο θέμα αυτών των συνταξιδοτικών μεταρρυθμίσεων. Και υπάρχει συνένεση πως χρειάζεται συντονισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως επίσης και ευρωπαϊκοί κανόνες για τα διασυνοριακά θέματα. Τα τελευταία δεκαετία αυτή τη στιγμή ο συντονισμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί ε, ο λίθο στον οποίο βασίζεται κάποιες προσπάθειες μεταρρύθμισης που λαμβάνουν υπόψη τη δημογραφική αλλαγή, την πίεση των αγορών, όπως επίσης και της αλλαγής του ρόλου των φύλων στην αγορά εργασίας. Πάντως κάποιοι ξεκίνησαν, κάποιοι προχώρησαν στις συνταξιδοτικές μεταρρυθμίσεις και κάποιοι ακόμα το σκέφτονται. Αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω πως για την έκθεση που διάβασα θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια γιατί στηρίζει απόλυτα αυτή την ολιστική προσέγγιση την οποία και εμείς προτιμήσαμε. Σε αρκετά σημεία φωτίζει ε, την ανάγκη βιωσιμότητας και τη σχέση με την ασφάλεια αυτή τη επάρκεια και βιωσιμότητα, όπω επίση εντοπίζει που υπάρχει ευρωπαϊκή προστιθέμενη εξουσία. Εμεί αυτή τη στιγμή ε, τελειώνουμε με τη διαδικασία αξιολόγηση τη διαβούλευση και θα λάβουμε υπόψη και τη γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεδομένου ότι η κατάσταση πιέζει, ήδη ετοιμαζόμαστε για τη λευκή βίβλο, την οποία θα παρουσιάσουμε στο ε, τρίτο τρίμηνο του 2011 να κλείσω λέγοντας πως μία από τις μεγάλες επιτυχίες του κοινωνικού μοντέλου της Ευρώπης είναι πως εξασφαλίζει πως η, η μεγάλη ηλικία, το γύρας δεν αποτελεί συνώνυμο της φτώχειας. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε και να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη να λάβουν τις σωστές αποφάσεις έτσι ώστε τα συνταξιδετικά συστήματα να ανταποκριθούν σε αυτούς τους στόχους. Τους τελευταίους μήνες έγινε πολύ έντονη και ζωντανή συζήτηση στον χώρο της συνταξιδοτικής μεταρρύθμισης και νομίζω πως η φετινή χρονιά θα είναι είναι εξίσου έντονη. Ε, θα ήθελα λοιπόν να στηριχθώ ε, σε εσά ε, έτσι ώστε να γίνει μια πραγματική αλλαγή για να έχουμε πραγματικά επαρκή ε, και βιώσιμα συστήματα συνδοξιδετικά στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε εκ μέρους της Επιτροπής Οικονομικών και Κοινωνικών Θεμάτων, κ. σκούτας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μιλάμε σήμερα στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου στα θέματα συνταξιωτικού συστήματος, που βέβαια είναι ευρωπαϊκή σημασία. Η γύρανση του πληθυσμού, η χρηματοοικονομική κρίση, η καθυστέρηση εισόδου των νέων στην αγορά εργασίας, όλα αυτά απαιτούν κοινή εργασία. Η αρχή της επικουρικότητας και τα εθνικά καθεστώτα είναι εκείνα, τα οποία καθορίζουν τα όρια στην ευρωπαϊκή παρέμβαση. όμω αν τα κράτη-μέλη εφαρμόσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα έχουμε πολύ καλύτερη λειτουργία τη ενιαία αγορά και θα μπορούμε να ενθαρρύνουμε την κινητικότητα των εργαζομένων. Προκειμένου τα δημόσια συστήματα συνταξιοδότηση να είναι αηφόρα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να παραμένουν στην αγορά εργασία μέχρι τη στιγμή τη συνταξιοδότησή του. Η αύξηση της ανεργίας είναι ένα φαινόμενο εξαιρετικά ανησυχητικό και επικίνδυνο. Η μεταρρύθμιση των συνταξιδοτικών συστημάτων λοιπόν θα πρέπει να συνοδεύεται με πολιτικές προαγωγής της εργασίας. Η μεταρρύθμιση των συνταξιδοτικών συστημάτων δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την... Θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με την φτώχεια χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικών στρωμάτων. Θα πρέπει τα κράτη να μπορούν να δίνουν κατάλληλα εισοδήματα, κατάλληλα εισοδήματα και επίπεδα συντάξεων για όλους τους εργαζομένους. Μέχρι στιγμής έχουμε προωθήσει την ιδέα μιας ευρωπαϊκής σύνταξης. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να μπορούν να εγγυηθούν ένα ελάχιστο σύνταξη, αλλά αυτό δεν είναι παρκές. Νομίζω ότι τα κράτη-μέλη μπορεί ενδεχομένως να είναι απρόθυμα να αφήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να εμπλακεί σε ένα πεδίο που είναι τη δική του κυριαρχία και αρμοδιότητα. Όμω παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για το επίπεδο ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Γιατί η κοινωνική δυστημία μπορεί να πυροδοτήσει πραγματικά εκπληκτικά φαινόμενα. Εάν σκεφτούμε τα προβλήματα πληθυσμών που πολύ συχνά θυσιάζονται προς το συμφέρον κρατών που δεν ενδιαφέρονται καθόλου για την ευημερία των πολιτών τους. Ευχαριστούμε κύριε Ντεγιόνκα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την μου για την καλή συνεργασία. Πράγματι συμπεριέλαβε πάρα πολλά από αυτά τα οποία είπε η Επιτροπή μας. Επίσης ε, Συμφωνώ ιδιαίτερα με αυτό το οποίο είπε πως ο καθένας θα πρέπει να ξέρει ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεται πώς διαμορφώνεται η σύνταξή του. Τώρα υπάρχει βεβαίως μια διαφορά μεταξύ των δηλώσεων της κυρίας Σόμεν Ρόιτεν και το εάν θα γίνει η συνταξιοδοτική πολιτική μέρος της ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης. Δεν θέλω εδώ πέρα να δημιουργηθεί εντύπωση πως ε, πηγαίνουμε προς μια αναθεώρηση των εθνικών αρμοδιοτήτων στο σημείο αυτό. Επίσης, οι προσπάθειες οι οποίες ε, γίνονται αυτή τη στιγμή να συνδεθεί η ηλικία συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο ζωής με ανησυχούν πάρα πολύ. Ειδικά για την Ολλανδία δεν νομίζω να χρειάζεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Από την Επιτροπή Γυναικών, η κυρία Ματερά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ την εισηγήτρια. Η προσοχή η πολύ μεγάλη που γίνεται στα πλαίσια τη πράσινη βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά το μέλλον των εξωτερικών συστημάτων στην Ευρώπη προκαλεί πραγματικά ανησυχίε. Υπάρχει αρνητική διάκριση εναντίον τη γυναίκες γιατί πιο συχνά διακόπτουν επαγγελματική σου προκειμένου να εξασφαλίσουν τη φροντίδα των παιδιών, των ε, άρρωστων μέλων τη οικογένεια και των ηλικιωμένων. Οι γυναίκες λοιπόν εκείνες οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη τάση σχέση με τους άνδρες να δεχθούν προσωρινές ε, ε, εργασίες ή απασχόληση ή μερικής απασχόλησης με επομένως με πολύ χαμηλότερη αμοιβή η οποία επομενω με πολυ χαμηλοτερη αμοιβη περίπου το 18% σε σχέση με τις ανδρικές αμοιβέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτή την αρνητική διάκριση λοιπόν οι γυναίκε καταλήγουν και σε πολύ χαμηλότερη σύνταξη σχέση με τους άνδρες, επιτείνοντας ε, τον ε, κίνδυνο ε, φτώχεια των ηλικιωμένων γυναικών, να λάβουμε υπόψη και το μεγαλύτερο προσδόκιμο ηλικία. Ή και ο χρόνος ο οποίο διαθέτουν οι γυναίκες στη φροντίδα παιδιών ή άλλων εξαρτώμενων μελών, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στο όλο σύστημα υπολογισμού της σύνταξης, μαζί με όλες τις άλλες συμβάσεις σχετικής εργασίας. Η Πράσινη Βίβλος έχει ανοίξει μια διαβούλευση. Ελπίζω λοιπόν στο ολο συστημα υπολογισμου της συνταξη μαζι με ολες τις αλλες συμβασεις σχετικη εργασια η πρασινη βιβλος εχει ανοιξει μια διαβουλευση ελπιζω λοιπον στο τελος του εσωτερικό, αν θέλετε, του νέας λευκής βίβλου να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή σε αυτά τα ευαίσθητα ζητήματα τη ακόμα μεγαλύτερη ανισότητα γυναικών και ανδρών σε ό,τι αφορά τον υπολογισμό των συνταξιδοτικών δικαιωμάτων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να πω και άλλα. Ναι, ίσως να, επι, να επιβάλλεται μια μικρή θετική διάκριση πέρα των γυναικών, λέει η Πρόεδρος. Και τώρα, ε, περνώ στους ε, αγορητές εκ μέρους των ομάδων. Καταρχάς για το, από το ΕΛΚΟ, κύριος Ορή. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός τροπολογιών, γύρω στις 500 έχουν υποβληθεί, το οποίο αποδεικνύει πως όλοι ενδιαφερόμαστε πάρα πολύ για το θέμα αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια γιατί τουλάχιστον ε, μας κίνησε την προσοχή, απλούστευσε την ε, κατάσταση έτσι ώστε να έχουμε ένα κείμενο το οποίο να αντικατοπτρίζει την τρέχουσα θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και όταν λέω τρέχουσα είναι γιατί αυτή τη στιγμή ξεκινά η συζήτηση για την Πράσινη Βίβλο, αναμένουμε και την Λευκή Βίβλο, οπότε βρισκόμαστε σε ένα πολύ αρχικό στάδιο των συζητήσεών μας. Συμφωνούμε βέβαια για τη διαφοροποίηση με τα όσα λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα ήθελα όμως να συμπιστώ την προσοχή και στο εξή. Υπάρχει χώρος για να είμαστε πιο ακριβείς στα όσα μιλάμε. Όταν μιλάμε λοιπόν για επικουρικά ταμεία, νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να ληφθούν δεόντως υπόψη. Και όσο για τη σταθερότητα, για τη σταθερότητα ίσως αυτήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και ε, που δεν είναι να θίξουμε την ασφάλεια των συνταξιδοτικών συστημάτων. Τα συνταξιδοτικά συστήματα δεν μπορούν ε, να λυθούν με συντονισμό μόνο σε θέματα συνταξιδότηση. Χρειάζεται περισσότερη οικονομική συνεργασία και ποιο θα πρέπει να είναι, ποιος θα πρέπει να είναι ο στόχος μας να εξασφαλίσουμε πως οι, οι ιδέες μας θα ε, συνδυάζονται και με τα όσα έχουμε στην στρατηγική για το 2020 που και την οικονομική διακυβέρνηση. Ο κύριος Νταρντέν για δύο λεπτά έχει το λόγο. Merci, Madame la Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιθυμώ καταρχά να, να υπογραμμίσω την πολύ σημαντική εργασία και τη συνένεση που απέτυχε η συγγήτρια. Συγχαρητήρια λοιπόν, Γεια. Σε οι συζήτησεις που οδήγησαν σε συμβασμό, οδήγησαν στην ε, καταπλειοψηφία υιοθέτηση του σχεδίου, ε, του σχεδίου της έκθεσης αυτής στην Επιτροπή Απασχόλησης κατά πλειοψηφία υπερψήφιση, ακριβώ ουσιαστικά είναι και μια υπερψήφιση προ του θεσμού. Η έκθεση αυτή για το μέλλον των συγκριτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι το μόνο ευρωπαϊκό θεσμικό ε, κείμενο αυτή τη στιγμή απέναντι στην ε, ετήσια έκθεση που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο σχετικό έγγραφο του ντουέτου Σαρκοζή Μέρκελ σε ό,τι αφορά τον αντίκτυπο τη ανταγωνιστικότητα. Το έγγραφο αυτό θέτει, αν θέλετε, και αμφισβητεί τον πρώτο πυλώνα και μια αυτόματη παράταση του τα αξιοδότηση. Ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο σχέδιο έκθεση, όπω έχει υιοθετηθεί, ουσιαστικά εκφράζεται για το θεμελιώδη ρόλο του πρώτου πυλώνα, που είναι ο θεματοφύλακα τη ε, βασική ε, σύνταξη, και η του δεύτερου πυλώνα για μια γενικευμένη επικουρική σύνταξη. Σε ό,τι αφορά την παράταση του χρόνου συνταξιοδότηση και παράταση του παραμονή στην αγορά εργασία περισσότερο παρά την ε, εξορισμού και μοιραία ε, επέκταση της, ε, του ορίου ταξιοδότησης. Ζητά έναν ενισχυμένο ρόλο των κοινωνικών εταίρων στον ορισμό και την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων των εξωτικών συστημάτων για την εξάλληψη των ανισοτήτων συντάξεων μεταξύ ανδρών και γυναικών που συνδέονται με από τις διακρίσεις όπως υπενθύμησε η Μπάρμπαρα. Με τα στοιχεία αυτά, με αυτά τα προοδευτικά στοιχεία και άλλα κόμμα που θέλω να τονίσω, χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να στείλει σαφές μήνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κοινωνικό και προοδευτικό κίνημα, ε, μήνυμα που ελπίζω ότι θα λάβει υπόψη για την μελλοντική σύνταξη της Λευκής Βίβλου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ντάγνα και τώρα τον λόγο έχει η κυρία Χάρκιν για τους ελεύθερους. Ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ. Θα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που με διευκόλυνε και να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση, η οποία πραγματικά είναι επίκαιρη. Κάποιοι μιλάνε για ορολογιακή βόμβα ε, και έτσι χαρακτηρίζουν το συνταξιοδοτικό. Γιατί βέβαια θα πρέπει να δούμε ποια είναι η διαφορά μεταξύ των όσων αποταμιεύουμε για τι ιδιωτικέ, δηλαδή επικουρικέ συντάξει και τι βασικέ συντάξει και την αυξημένη ανάγκη κονδυλίων για να εξασφαλίσουμε τη συντάξη τα επόμενα 40 χρόνια. Αυτό λοιπόν το έλλειμμα είναι τεράστιο, άρα ο χαρακτηρισμός ως ορολογιακή βόμβα είναι σωστός. Χρειάζεται λοιπόν με κάποιο τρόπο να αφοπλίσουμε αυτή την ορολογιακή βόμβα. Αυτή είναι η διαδικασία η οποία τρέχει τώρα, αλλά το ερώτημα κλειδί είναι ποιο είναι υπεύθυνο. Νομίζω ότι είναι τα κράτη-μέλη τα οποία έχουν την ευθύνη να εξασφαλίσουν πω υπάρχουν επαρκεί συντάξει για του πολίτε του. Όμω Ξέρουμε πως οι οικονομίες αυτή τη στιγμή των κρατών μελών βρίσκονται σε αλληλεξάρτηση. Οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες συντονισμού που έχουμε. Δεν νομίζω πάντως πως γίνεται αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει όρια σύνταξης ή συνταξιδοτική ηλικία. Θεωρούμε πάντως πως τα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ορίσουν την επάρκεια που είναι ε, το να ζουν με αξιοπρέπεια ηλικιωμένοι. Χαίρομαι λοιπόν που επίσης τονίσαμε την πτυχή, ε, την πτυχή του φύλου και νομίζω πως θα πρέπει να δούμε και την κινητικότητα όπως επίσης και την στρατηγική για το 2020. Τέλος, στηρίζω το γεγονός πως θα πρέπει στο ε, Ίσπα αυτή τη στιγμή να ε, ενταχθεί το θέμα τη ε, της εξασφάλισης κονδυλίων για τις συντάξεις. Δεν μπορούμε το θέμα αυτό να το αφήσουμε στην άκρη. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ ε, για δύο λεπτά. Το, κυρία Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να προσθέσω τη φωνή μου σε όσους ευχαρίστησαν την εισηγήτρια για την πολύ καλή δουλειά της στην έκθεση αυτή, γιατί όλοι γνωρίζουμε πως υπάρχουν εθνικές διαφορές, διαφορές μεταξύ των πολιτικών ομάδων μας και το να καταλήξουμε σε κάτι το οποίο θα βρει στήριξη είναι κατόρθωμα. Η ομάδα μου είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένη για το ότι η έκθεση αυτή αναγνωρίζει την σημασία των συντάξεων του πρώτου πυλώνα. Η δέσμευση για ένα επαρκές επίπεδο το θέμα το του πώς θα μπορέσουν να διασφαλίσουν μια αξιοπρεπή ζωή. Γιατί βεβαίως μην ξεχνάτε πως ε, το 2010 ασχοληθήκαμε με ζητήματα φτώχειας και βεβαίως ένα σταθερό εισόδημα για όλους είναι μια ουσιαστική εγγύηση. Και θα, επίσης θα ήθελα να καλωσορίσω την αναγνώριση του ότι πρέπει να δούμε τις επαρκείς συντάξεις για τις γυναίκες. Επίσης αναγνωρίζουμε την σημασία της αντιμετώπισης ε, Τη διάκριση που υφίστανται οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι και να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να μείνουν στη δουλειά. Για εμά. επίσης, ε, το να μπορούν να μεταφέρονται τα συνταξιδοτικά δικαιώματα είναι κάτι το σημαντικό όλο και περισσότερο. Οι άνθρωποι δεν εργάζονται για μία εταιρεία σε ολόκληρη τη ζωή τους, εργάζονται για πολλέ και όχι πάντα στην ίδια χώρα. Και πρέπει να αποφύγουμε αυτό τον κατακαιρματισμό τη παροχή συντάξεων. Οπότε υπάρχει ένα ουσιώδη ρόλος εδώ πέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, είμαστε ικανοποιημένοι για το ότι η έκθεση αυτή περιέχει μια δέσμευση για την παροχή του δεύτερου πυλώνα που θα πρέπει να είναι διαθέσιμος χωρίς ε, διάκριση για λόγους ε, ηλικίας, ε, φύλου ή μορφής εργασίας, εργασιακής σχέσης. Επίσης είμαστε ικανοποιημένοι ούτως ή άλλως από το ότι η Κομισιόν αντιμετωπίζει το πράγμα ε, από πλευράς κύκλου ζωή και βεβαίω με ό,τι αυτό σημαίνει θετικό και αρνητικό και αναγνωρίζουμε τη σημασία της αλληλεγγύης στον πρώτο πυλώνα και για αυτού ε, οι οποίοι βρίσκονται ίσως ε, σε μια σχέση αποσχόληση που είναι πιο ευκαιριακή με βραχυχρόνια συμβόλαια κτλ. Επίσης, για τον τρίτο πυλώνα, τον ιδιωτικό, είναι σημαντικό εάν οι άνθρωποι το επιλέγουν να έχουν επαρκείς και πλήρεις ε, πληροφορίες. Επίσης καλωσορίζουμε το ότι ε, αυτό το οποίο λέει η έκθεση, αν δηλαδή είναι να υπάρξουν αλλαγέ στι συνταξιωτικέ διατάξει, θα πρέπει να υπάρχει επαρκή χρόνο για να επανεξετάσουν οι άνθρωποι το οικονομικό του μέλλον. Ευχαριστώ, κυρία Λάμπερτ, η κυρία Γκίρλινγκ. Έχει τώρα τον λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ομάδα μου υποστηρίζει τη δημοσίευση αυτής της πράσινης βίβλου. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη και έρχεται ακριβώς σε μια στιγμή όπου γίνεται συζήτηση σε όλα τα κράτη-μέλη των θεμάτων που αναφέρθηκαν πριν. Ε, όχι μόνο τη απασχόληση, αλλά και τη αλλαγή της δημογραφικής, πολύ μεγάλης πρόκλησης ε, μεταξύ των κοινωνικών φύλων και το καθεξής. Η έκθεση αυτή αναγνωρίζει τη σημασία του να μοιραστούν τι βέλτιστε πρακτικέ μεταξύ, μεταξύ τους κράτη-μέλη, να υπάρξει ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά τονίζει επίση ότι παραμένει τη αρμοδιότητα του κράτου μέλους στο θέμα τη σύνταξη. Αναγνωρίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να θεσμοθετήσει ούτε σε ό,τι αφορά τι ηλικίε ταξιοδότησης, ούτε το επίπεδο των συντάξεων. Ζητά όμω με σαφήνεια και κατηγορηματικά πραγματικότητα να υπάρχει διευθέτηση στα κράτη-μέλη σε συνάρτηση και λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις συνθήκες κάθε κράτος μέλος. Πιστεύω ότι είναι θεμελιώδη σημασία η περαιτέρω δουλειά για την μεταφορά και τη δυνατότητα μεταφορά εξωτερικών δικαιωμάτων. Γιατί ακριβώ υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα και έχω συναντήσει πάρα πολλού ευρωπαίου πολίτε οι οποίοι κινούνται για λόγου δουλειά σε διάφορα κράτη και δεν πρέπει να παγώνουν τα εξωτερικά του δικαιώματα οι προσδοκίε αλλάζουν. Αλλάζουν δημογραφικά στοιχεία, αλλάζουν και οι προσδοκίε. Και πρέπει και είναι απαραίτητο να μπορούμε να συντονιστούμε και στην εκπόνηση πολιτικών σχέση με τι αλλαγέ αυτέ που αλλάζουν. Ευχαριστούμε κυρία Φιγκερέιντο για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε ότι υπάρχει μια πρόταση που είναι ακριβώς το σύμφωνο ανταγωνιστικότητα. Το διευθυντήριο, το οποίο διοικείται από τη Γερμανία, προσπαθεί να πλήξει ακόμα περισσότερο το καθολικά θεσπισμένο δικαίωμα της κοινωνικής ασφάλισης, αυξάνοντας το όριο αξιοδότηση, μειώνοντας τους μισθού και μαθημοποιώντα τι συντάξει αυτέ με ρυθμό με, τον, ε, με το ποσοστό πληθωρισμού, το οποίο βέβαια είναι προ όφελο του ευρύτερου χρηματοοικονομικού τομέα που ξέρετε ότι θέλει να έχει περαιτέρω κερδοσκοπικά κέρδη, χάνει τη χρηματοδότηση και ιδιωτικοποίηση των ιδιωτικών συστημάτων. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι δρόμο παίρνει η Ευρώπη που βασίζεται σε πολιτικές αντικοινωνικές και δυστυχώς ε, η έκθεση αυτή οδηγεί αυτό τον, ε, με αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ της λόγω έκθεσης με σύνδεση που γίνεται μεταξύ του προσδόκιμου ηλικία και μιας πολύ πιο παραεταμένης διάρκειας ε, εργασίας, χώρων εργασίας. Και γίνεται λόγος επίσης το έγγραφο αυτό για παρέμβαση του ιδιωτικού τομέα, ενώ ξέρουμε ότι υπάρχουν πολύ σοβαροί κίνδυνοι σε ό,τι αφορά τις κερδοσκοπικές τάσεις και εκμετάλλευση των ε, ταμείων. Γιατί βλέπουμε πάρα πολλές γυναίκες συνταξιούχους να βρίσκονται σε πολύ φτώχεια λόγω αυτής της κερδοσκοπίας. Χρειάζεται λοιπόν να τροποποιηθεί το συνταξιωτικό σύστημα χωρίς όμως να ρίξουμε το επίπεδό του. Θα πρέπει να υπάρχει ένα συγκεκριμένο δικαίωμα δεδομένο για όλους τους νέους, να υπάρχει μεγάλη, κάποια αφορολόγηση σε ό,τι αφορά τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές και τις χρηματιστηριακές ε, πράξεις και να είμαστε κατά της περαιτέρω αύξησης του ορίστου αξιοδότηση. Και θα πρέπει να υπάρχει ένα καθολικό και δημόσιο σύστημα ε, αξιοδοτικό στήματο. Θα πρέπει να υπάρχει μια μεταρρύθμιση που θα σέβεται τους ηλικιωμένου και θα του επιτρέπει να ζουν με αξιοπρέπεια και με τους στόχους που είχαν ε, τεθεί από την αρχή, δηλαδή την εξάλληψη τη της φτώχειας. Αυτό ισχύει για τη Γαλλία, την Ελλάδα και όλες τις άλλες χώρες. Ευχαριστούμε κύριο Κλάρκ για ένα λεπτό. Στην Επιτροπή Απασχόλησης πέρσι 22 Νοεμβρίου είπε η συγγήτρια πως η συντάξη είναι αποκλειστική αρμοδιότητα των κρατών μελών. Και τώρα μας λέει, παρά το ότι παίζουν ηγετικό ρόλο, υπάρχουν πτυχές συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην παράγραφο 9 η πράσινη βίβλος τονίζει την αρμοδιότητα των κρατών μελών, αλλά τα καλεί να συντονίσουν τις πολιτικές της. Εδώ πέρα έχουμε διγλωσία. Η Εθνική Ένωση Συνταξιδοτικών Ταμείων του Ηνωμένου Βασιλείου λέει πως ε, σύμφωνα με αναλογιστικές μελέτες θα γίνουν πιο ακριβές κατά 90% συντάξει. Έστω και αν αυτό το ποσό είναι υπερβολικό, σημαίνει πως θα χρειαστούν πάρα πολλά ποσά και βεβαίως θα αυξηθούν τα ασφάλιστρα. Οι συνταξιδοτικέ εταιρείε και τα κράτη-μέλη δεν χρειάζονται αυτή την έκθεση, χρειάζονται βοήθεια για να κρατήσουν τα ασφάλιστρα χαμηλά. Αλλιώ αυτή η έκθεση έχει την δυνατότητα να καταστρέψει αυτό το οποίο θέλει να προστατεύσει. Τον λόγο έχει η κυρία Λεπέν για ένα μισή λεπτό. Ε, αγαπητοί συνάδελφοι, στην Ευρώπη του Συμφώνου Σταθερότητα και αύριο του Συμφώνου Ανταγωνιστικότητα, η μεταρρύθμιση των σχετικών συστημάτων ε, είναι στο στόχο. Πώ μπορεί να υπάρξει ανταγωνιστική Ευρώπη αν αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη που έχουν έλλειμμα πρέπει να είναι σε απόλυτη ισορροπία μέχρι το 2013. Η απάντηση είναι να παρατείνουν τον χρόνο συνταξιότητα του 27ο και να υπάρχει μια ριζική μεταρρύθμιση κατά τμήματα ώστε να μειωθούν τα συλλογικά δικαιώματα και παροχέ οι πολιτέ δεν αυταπατώνται γιατί ζητάτε ένα εγγυημένο ακατόφλι χαμηλότερο επίπεδο αν θέλετε σύνταξη και το οποίο μα ζητείτε να δίνουμε και στου ξένου που έχουν φτάσει εδώ και ποτέ δεν έχουν καταβάλει καμία εισφορά. Εξάλλου, η έκθεση αυτή θα αυξήσει ακόμα περισσότερο την πίεση στα κράτη-μέλη και να τα οθήσει να αναπτύξουν προγράμματα σταξιοδότηση κεφαλαιοποιητικά, των οποίων γνωρίζουμε του προφανεί μείζονε κινδύνου που παρουσιάζουν. Είπαμε ότι τα σχετικά συστήματα είναι τη αρμοδιότητα των κρατών μελών. Όμω, εναντίον τη θέληση των λαών, αυτή τη στιγμή θέλουμε να βάλουμε μια δημοσιονομική πειθαρχία άνευ προηγουμένου. Και όντω έτσι είναι. Οι, οι υπάλληλοι, αν θέλετε, οι ευρώ οι υπάλληλοι, αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να σώσουν μια υπερφιλελεύθερη Ευρώπη ει βάρο των γενικών πολιτών. Ευχαριστούμε στου μη γεγραμμένου τώρα. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Είναι καλό το ότι μία έκθεση πρωτοβουλίας δεν κρύβεται την Δευτέρα για να την ξεπετάξουμε. Και ο λόγος βεβαίως είναι ακριβώς οι πάρα πολλές αυτές τροπολογίες γύρω στις 500 και από τις δύο επιτροπές. Ξέρετε πως στην Γερμανία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία και Αυστρία δυστυχώς αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία να, να εφαρμοστούν νέες ελάχιστες προδιαγραφές για τι ε, συντάξει και το κομμάτι του εκείνο το οποίο καταβάλλεται από τι επιχειρήσει, Κάτι το οποίο βεβαίω σημαίνει μια αύξηση του κόστου έω και 40%. Και βεβαίω αυτό το οποίο έγινε από του κοινωνικού εταίρους δεν μπορεί να καταργηθεί. Επίση, λήφθη απόφαση πως ε, θα πρέπει όλες οι ελάχιστες απαιτήσει της οδηγίας ε, φερεγγιότητα 2 να ισχύσουν και για τα συνταξιδοτικά ταμεία. Βεβαίως αυτό είναι βήμα προόδου αν και δεν αποτελεί εγγύηση για τα προϋπάρχοντα συνταξιδοτικά ταμεία. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει ένας ορισμός για την επάρκεια των συντάξεων και βεβαίως δεν έγινε δεκτό το να έχουμε μια ενιαία ηλικία σύνταξιοδότηση ε, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δικαίωση, οι κύριοι Σαρκοζή και Μέρκελ ε, είπαν πως πρέπει να έχουμε μια σταδιακή προσέγγιση γιατί υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής και τα δημογραφικά στοιχεία. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τις ε, διατάξεις αυτές καθώς εδώ πέρα οι κρεμότητες οι οποίες υπάρχουν είναι μεγαλύτερες από αυτές οι οποίες καλύπτονται από την σωτηρία από την ομπρέλα σωτηρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εισηγήτρια ήθελε να σας κάνει μια ερώτηση. Το δέχεστε? Παρακαλώ, κυρία μου. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να αιωρούνται πράγματα εδώ μέσα. Γι' αυτό θέλω να μας πει ο κύριος Μαν που βρίσκεται σε αυτή την έκθεση πως θα πρέπει να προσαρμοστεί ε, η οδηγία φερεγγιότητας στον δεύτερο πυλώνα. Εγώ, είμαι κατά, αλλά που, ε, εγώ δεν είμαι κατά, αλλά πού το αναφέρει. Θέλετε να απαντήσετε στην εισηγήτρια, παρακαλώ. Είχαμε δύο εκθέσεις από δύο επιτροπές. Εκεί πέρα υπάρχει η σύσταση να εφαρμοστεί η οδηγία φερεγγιότητας δία στα συστήματα επιχειρηματικής ε, σύνταξης. Είχαμε τέτοια εμπειρία στη Γαλλία. Σε άλλες χώρες δεν υπάρχει αυτή η εμπειρία. Πρέπει να το δούμε σε πολύ μεγάλη λεπτομέρεια το ζήτημα. Από μια λευκή βίβλο να πει, προσπαθήστε να πείστε τους άλλους που δεν έχουν την εμπειρία στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Οπότε νομίζω μπορούμε να το εξετάσουμε. Μπήκαμε λοιπόν στις λεπτομέρειες. Η κυρία Μπερές έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Επίτροπε, η συζήτηση αυτή είναι η συζήτηση προσανατολισμού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέλει να σας στείλει ένα μήνυμα. Όμως η ζωή αλλάζει. Το θέμα το συνταξιδοτικό το έχουν θίξει σε άλλα βήματα. Ίσως λοιπόν σε αυτό το σύμφωνο σταθερότητας και στο σύμφωνο ανταγωνιστικότητας πείτε μου τι θα κάνετε με το όριο συνταξιδότησης που προτείνεται να είναι τα 70 έτη η, Ευρωπαϊκή, κοινωνική Ευρώπη νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό οικοδομείται εναντίον των λαών της και δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Τώρα η συγγήτρια μας είπε πως υπάρχουν πολλά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Εγώ λοιπόν σας παρακαλώ τη στιγμή που θα ετοιμάσετε τη θέση της Κομισιόν για την Λευκή Βίβλο να τα λάβετε υπόψη και να αναγνωρίσετε πως υπάρχει για παράδειγμα το θέμα του φύλου το οποίο κατά τη γνώμη μας δεν εξερευνήσατε επαρκώς. Επίσης Είπατε πως ο καλύτερος τρόπος να ρυθμίσετε το θόμα των ε, συντάξεων είναι να προκρίνετε την απασχόληση. Και αντί να λέμε ποια θα είναι η νόμιμη ηλικία ε, συνταξιοδότηση, να λέμε ποια θα είναι η πραγματική. Όμως η έκθεση συγγήτριας για μας, τους Γάλλους σοσιαλιστές, έχει συμπεριλάβει μια ένδειξη η οποία είναι προβληματική και για την οποία δεν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή την ιδέα πως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής θα πρέπει να αναπροσαρμόσει αυτόματα το όριο ηλικία συνταξιοδότησης προς τα επάνω. Νομίζω πως με τον τρόπο αυτό οπισθοχωρούν τα κοινωνικά δικαιώματα. Και θα ήθελα τέλος να πω πως χωρίς ε, κοινωνικό διάλογο, χωρίς ε, να ε, λάβουμε υπόψη τη γνώμη των κοινωνικών εταίρων, δεν θα φτάσουμε πουθενά. Θα είναι σαν να προσπαθήσουμε να χτυπήσουμε πάνω σε ένα τείχο. Ευχαριστώ πολύ. Ε, κύριο Στέρξ, ευχαριστώ. Θεωρώ πως η συγκήτρια βρήκε πολλές ισορροπημένες απαντήσεις ε, σε τα ερωτήματα της Κομισιόν. Κοιτάξτε, όταν τονίζουμε βεβαίω την σημασία του πρώτου πυλώνα, δικαίως πρέπει να δούμε πως ε, είναι εξίσου σημαντική η κατάσταση των δημοσίων οικονομικών που στηρίζουν τον ε, πρώτο πυλώνα. Οπότε πρέπει να δούμε ποια βάρη, συνταξιοδοτικά βάρη, έχει το κράτος ε, μακροπρόθεσμα και είναι σε θέση να σηκώσει. Οπότε η Κομισιόν θα πρέπει να αναλάβει μία μελέτη για να δούμε πού βρίσκονται οι κίνδυνοι και οι δυσκολίες. Δεύτερον, θεωρώ πως και στον δεύτερο πυλώνα θα πρέπει ε, να παίξει ένα ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ πέρα βέβαιως παίζει ρόλο η φερεγγιότητα 2 να δει η Κομισιόν ποιο είναι μακροπρόθεσμα ο κίνδυνο και να ξεκαθαρίσει πώ θα πρέπει να καλυφθεί αυτό ο κίνδυνος και να δούμε συγκεκριμένα μακροπρόθεσμα γενικά για τα συνταξιοδοτικά συστήματα ποιο είναι ο κίνδυνος, όχι ενό είδου για όλων των ειδών τα συνταξιοδοτικά συστήματα. Γιατί όπω και η κυρία Χάρκιν φοβούμαι και εγώ πω δεν έχουμε αντιληφθεί ποιοι είναι οι κίνδυνοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ κύριο Σιμάνσκι για ένα λεπτό. E, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Το σχέδιο ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πραγματεύεται σε, όλη, σε όλες που έγινε εδώ στο Κοινοβούλιο, που συζητήθηκε. Συνιστά την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών και συζητά το πόσο ευάλωτα είναι ακόμα τα συνταξιωτικά συστήματα. Στα πλαίσια τη της συζήτηση στην Επιτροπή Απασχόληση υπογραμμίσαμε την πολύ μεγάλη σημασία των δημογραφικών αλλαγών για τη μελλοντική μορφή των συνταξιωτικών συστημάτων. Είναι σημαντικό λοιπόν να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αντιμετωπιστεί η δημογραφική κρίση στην Ευρώπη. Αξιολογώντα ταυτόχρονα τα συλλογικά συστήματα, αναφέρεται σε συμπεράσματα ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι πολύ μεγάλε διαφορέ που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών και σε ό,τι αφορά τις ε, ε, δυνατότητες χρηματοδότησης συστημάτων, αλλά και στο πεδίο των υφιστάμενων ε, συστημάτων στις χώρες αυτές. Ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Χάντελ για ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, η ευημερία της κάθε χώρας είναι η αξία που δημιουργούν οι άνθρωποι με την εργασία τους. Γι' αυτό θα πρέπει και η κοινωνική εργασία να μετρήσει. Οι άνθρωποι θα πρέπει βεβαίως στην τρίτη ηλικία να απολαμβάνουν μια κάποιε φροντίδα. Αλλά η κρίση κατέδειξε πω ε, μόνο οι δημόσιε συντάξει είναι αξιόπιστε. Αντιθέτω, ε, οι επιχειρηματικές και ιδιωτικέ συντάξει ε, έχουν και αποδείχθηκε αυτό στην ε, κρίση μισή κινδύνου κατά εκατομμύρια φορέ μεγαλύτερε από, αυτές, ε, από αυτού του οποίου μπορούν να καλύψουν. Και είναι παράλογο να λέμε πω έτσι θα καλύψουμε τι συντάξει. Οι άνθρωποι πληρώσανε και μια ομπρέλα για τις μεγάλες ε, τράπεζες και τώρα πληρώνουν με ε, λιτότητα και τώρα θα πρέπει να πληρώσουν και πάλι με μειώσεις των συντάξεων και οι τωρινές ε, οι μεταρρυθμίσεις οδηγούν σε αύξηση της φτώχειας. Άρα θα πρέπει εδώ πέρα να ενισχύσουμε τις σίγουρες δημόσιες συντάξεις και συνταξιωτικά συστήματα. Ευχαριστώ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Προσεχώς θα αντιστραφεί η ηλικιακή πυρημίδα στην ε, Ευρώπη. Οι 55χρονοι θα αποτελούν τη μεγαλύτερη ε, μερίδα του πληθυσμού και οι νέοι θα μπαίνουν όλο και πιο αργά στην αγορά εργασίας. Τα αποτελέσματα τα γνωρίζουμε όλο, θα έχουμε όλο και μεγαλύτερα διεύσοδα όσον αφορά τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι μια πολιτική φιλική προς την οικογένεια στην Ευρώπη είτε αφορά την φορολογία του οικογενειακού εισοδήματος είτε στον κοινωνικό τομέα για να υπάρξει αυτό το σύμφωνο των γενεών για να μπορέσουμε να δούμε πώς θα μειωθούν οι εισφορές ε, που πληρώνει μια οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν να δημιουργηθούν κίνητρα για να παραμείνουν ε, και ηλικιωμένοι περισσότερο στην εργασία. Και εδώ πέρα θα ήθελα να πω κάτι στον ε, κύριο Επίτροπο. Η μαζική μετανάστευση την οποία λέτε είναι ο λάθος τρόπος για να διασφαλίσουμε τις ε, συντάξεις μας και διακινδυνεύει και την κοινωνική ειρήνη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιάσλο Βιέτσκα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτές οι αλλαγές, οι δημογραφικές, η μείωση των γεννήσεων, τα διάφορα προνόμια τα οποία παρέχουν τα συνταξιδετικά συστήματα, όλα αυτά αποτελούν τεράστια πίεση για ε, τους ε, κρατικούς προϋπολογισμούς. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν σε ποιο βαθμό τα τρέχοντα συνταξιδοτικά συστήματα μπορούν να εξασφαλιστούν πρώτον και κατά πόσο μπορούν να εξασφαλίσουν και ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Νομίζω όμως πως αυτό αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών. Μιλάμε για διαδικασίες εξαιρετικά δαπανηρές, ε, μακρόχρονες και εδώ θα πρέπει να αποφασίσουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μαζί με το Συμβούλιο για να δούνε πώς μπορούν αυτό το επιπλέον κόστος να ληφθεί υπόψη από τα κράτη-μέλη. Οποιαδήποτε άλλη λύση θα μας οδηγήσει σε μια κατάσταση όπου τα κράτη-μέλη θα φοβούνται αυτό το επιπλέον ε, κόστος και δεν θα κάνουν το βήμα της μεταρρύθμισης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια του συνταξιδοτικού συστήματος, αλλά για να κάνουμε κάτι τέτοιο θα πρέπει να διαφοροποιήσουμε την πηγή ε, των κονδυλίων και να χρησιμοποιήσουμε και τα ε, κρατικά συνταξιδοτικά ταμεία αλλά και τα επικουρικά ιδιωτικά ταμεία. Αυτό θα εξασφαλίσει την σταθερότητα του συστήματος όπως επίσης και την ανάπτυξη της αγοράς εργασίας. Θα πρέπει επίσης να πούμε πως θα υπάρχει και μία νόμιμη εξωτερική ε, ηλικία που θα λαμβάνει υπόψη το γεγονός πως οι Ευρωπαίοι πια ζουν περισσότερα χρόνια. Χρειάζονται λοιπόν οι σωστές μεταρρυθμίσεις και στην αγορά εργασίας έτσι ώστε να υπάρχει κατάρτιση και συστήματα περίθαλψης για τους εργαζομένους. Σας ευχαριστώ κυρία μου λοιπόν για την βοήθειά σας και την συνεργασία σας. Ο κύριος Γκουτέρες Πριέτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Όλα το έχουν πει οι συνάδελφοι. Η σπονδυλική στήλη ε, των συνταξιδοτικών συστημάτων στην Ευρώπη είναι τα δημόσια συνταξιδοτικά συστήματα. Είναι τα μόνα που εξασφαλίζουν και τη συνοχή αλλά μειώνουν και τον κίνδυνο φτώχεια τη κοινωνία μα. Είναι εντυπωσιακό πω οι χώρε του ΩΣΑ αυτή τη στιγμή κάνουν τις μεγαλύτερες δαπάνες από τον προπολογισμό τους ε, στο, ε, στις συντάξεις. Και πρέπει να σας πω πως αυτή τη στιγμή τα συνταξιδοτικά ταμεία βρίσκονται πολύ μακριά από το όριο της φερεγγιότητας που έχουμε δεσπίσει. Θα πρέπει λοιπόν με εγκάρσιο τρόπο να ε, λύσουμε το πρόβλημα αυτό ε, της πίεσης με φιλόδοξες πολιτικές που θα ε, προωθήσουν τις γεννήσεις με διαφορετική πολιτική απασχόληση και ενδεχομένως και μεταναστευτική που θα εξασφαλίζει την ένταξη των μεταναστών έτσι ώστε να αντισταθούμε σε αυτές τις δημογραφικές πιέσεις και θα πρέπει να περιορίσουμε τις διάφορες τις διάφορες ε, απάτες που διαπιστώνουμε με τις εισφορές και τα λοιπά από τις εταιρείες. Γιατί αυτή τη στιγμή ζητάμε όλο και περισσότερο από τους εργαζόμενους ε, για να έχουν αξιοπρεπείς συντάξεις. Θα πρέπει να έχουν και αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας, λέω εγώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Λίν. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την πολύ σκληρή δουλειά που έχει κάνει δουλειά, για την έκθεση αυτή. Είναι εξαιρετική δουλειά τη. Καθίστε σαφέ ε, ότι οι συντάξει είναι πρωτίστω και κυρίω ε, αρμοδιότητα και ευθύνη των κρατών μελών. Ευτυχώ ε, απορρίψαμε οποιαδήποτε έκκληση για θέσπιση ελάχιστη σύνταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή για την εφαρμογή φερεγκαιότητα 2 στο θέμα των συντάξεων. Η συνθήκη τη Λισαβόνα το καθιστά σαφέ ότι η αρμοδιότητα συντάξεων δεν είναι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά των κρατών μελών. Αυτό όμω μπορούμε να κάνουμε να μοιραστούμε με τις βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες. Χαίρομαι που η τροπολογία μου η οποία ζητά την τροπολογία της ε, ε, οδηγίας απασχόληση 2000 ε, έχει επίσης συμπεριληφθεί και σε ό,τι αφορά ακριβώς το ηλικία ταξιοδότησης. Σε ό,τι αφορά το φιλοτικό όριο, το έλεγα πάντα ότι αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να κρατήσουμε σε επίπεδο κράτους κράτου μέλους το θέμα του, και του ασφαλίστρου και του ορίου ταξιοδότησης αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να διασφαλίσουμε την, να, να εξαλείψουμε την αναγκαστική σταξιοδότηση σε συνάρτηση με την ηλικία και να μπορούν να μείνουν άνθρωποι αν θέλουν στον χώρο εργασία. Ε, Δυστυχώ δεν υπάρχει αυτό στην έκθεση. Και τώρα ο κ. Κάβρον για ένα λεπτό. Εκτό μικροφώνου. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίε και κύριοι, Θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Ε, Αντιμετωπίζοντα τι εκατοντάδε τροπολογιών που κατατέθηκαν. Αν και δεν πρόκειται για νομοθετικού περιεχομένου έκθεση, είναι ύψιστη σημασία για την ε, <clears throat> βιωσιμότητα των εξωτικών συστημάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέλλον. Οι κυρίε αρχέ που λαμβάνει είναι Οι αποφάσει για τα εξωτικά συστήματα είναι πολιτικέ αποφάσει που είναι πλήρω και κατά αποκλειστικότητα ευθύνη των εγγονωμένων κρατών μελών είναι απαραίτητο να ε, παραταθεί, να αυξηθεί το όριο αξιοδότησης. Ο μόνος ε, πόρος ε, και πλούτου στην Ευρώπη στο μέλλον είναι η μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί η παραγωγικότητα και η απασχολησιμότητα όλων των εργαζομένων με μεγαλύτερη ευελιξία των εργασιακών σχέσεων και το σωστό μοντέλο εξωτικών συστημάτων που πρέπει να εισαχθεί. Δεν είναι σωστό να συντονιστούν τα συστήματα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν υποστηρίζουμε οποιαδήποτε προσπάθεια εναρμόνισης είτε ορίων ταξιοδότηση είτε σύνδεση ορίων ταξιοδότηση με το προσδόκιμο ηλικία. Δεν υποστηρίζουμε καμία ε, προσπάθεια για τον καθορισμό του ορισμού όπω το τι είναι επαρκή σύνταξη επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Λιωτά επικουρικότητα. Έχουμε επικουρικότητα, είναι η υπόθεση των κρατών μελών και πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα. Αυτό μα λέει συνέχεια η συγγήτρια. Εγώ θεωρώ πω η πράσινη αυτή βίβλος πρέπει να πάει κατευθείαν στα σκουπίδια. Και μάλιστα το κρίνει εδώ πέρα ως θετικό η συγγήτρια, γιατί επιμένει στην επικορικότητα από τη μία η, η συγγήτρια, από την άλλη, μας δίνει πάρα πολλούς ε, λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να ισχύσει κάτι τέτοιο. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ορίσει ελάχιστα ποσά. Πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αυξήσει την ηλικία σταξιδότηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προωθήσει τον ε, ανταγωνισμό μεταξύ των ταμείων και την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση. Ποια επικουρικότητα. Όλα αυτά ε, τουλάχιστον εάν οδηγούσαν σε μια πιο κοινωνική κατεύθυνση, να δεχόμασταν ότι έχει κάποιον ρόλο να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ πέρα όμως μόνο που θα μεγενθύνουμε το χάσμα μεταξύ πλουσίων και φτωχών. Ευχαριστώ. Τον, ρόλο, τον, λόγο τώρα έχει ο κύριος Κάζα για μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας την κυρία Όμεν Ρόιτεν για το εξαίρετο έργο της το έργο αυτό αναγνωρίζει, το, η έκθεση αυτή αναγνωρίζει το ότι σε μια εποχή στην οποία είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι οι Ευρωπαίοι πολίτες θα πρέπει τα κράτη-μέλη να διασφαλίσουν πως η κοινωνική προστασία και ειδικά τα συστήματα τα συνταξιοδοτικά είναι ισχυρά και θα μπορέσουν να δώσουν την βεβαιότητα στους Ευρωπαίους μιας οικονομικά ανεξάρτητης ζωής. Θα θέλουμε λοιπόν να τονίσουμε πως τα κράτη-μέλη πρέπει να ορίσουν την επάρκεια ως, ε, το, ως προς το τι είναι αναγκαίο για να ζήσουν αξιοπρεπώς οι ηλικιωμένοι. Αυτό βεβαίως πρέπει να καθοριστεί σύμφωνα με το τι ισχύει στο κάθε κράτος μέλος. Έξω και η αρχή της ε, επικορικότητας η οποία πρέπει να γίνει σεβαστή. Καλωσορίζω όμως ε, το ότι η Κομισιόν ε, ζητάει να υπάρξουν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Πρέπει λοιπόν για να επιτύχουμε τους στόχους οποίους έχουμε να υπάρξει μια μεταρρύθμιση για να υπάρχει βιωσιμότητα των συνταξιδοτικών συστημάτων, ειδικά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Και βεβαίω πρέπει να ληφθεί υπόψη το κόστος μεταρρύθμισης ακόμα και στο πλαίσιο της οικονομικής διακυβέρνησης. Ευχαριστώ κυρία Γκέντς για ένα λεπτό πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερο ευρωπαϊκό συντονισμό στα στεξιωτικά στήματα όσο είναι δυνατόν. Καταρχά, ε, είμαστε αντιμέτωποι μια κρίση που γύρει το ζήτημα τη μακροοικονομική σταθερότητα. και επίση γύρονται ζητήματα σχετικά με την ζωή των ε, πολιτών τρίτη ηλικία που πρέπει να διαβιούν με αξιοπρέπεια. Είδαμε ότι σε πάρα πολλέ χώρε δίνονται διαφορετικέ κατευθύνσεις στο πώ αναπτύσσονται τα διάφορα εξωτικά συστήματα. Ανεξαρτήτως των ελεγών που θα επέλθουν όμω, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει βιωσιμότητα αξιωτικών συστημάτων και ε, αξιοπρέπεια των ατόμων τρίτης ηλικία. Πρέπει να συζητήσουμε τα ζητήματα από του εταίρους, πρέπει να δώσουμε περισσότερους χρόνους, μεγαλύτερη μεταβατική περίοδο για την αλλαγή των συστημάτων, πρέπει να πληροφορήσουμε τους πολίτες πώς αλλάζουν τα πράγματα, θα πρέπει να μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις με πλήρη πληροφόρηση και θα πρέπει να αντιμετωπίζουν φιλικό τρόπο ανεξαρτήτως των αλλαγών. Ευχαριστούμε. Κυρία Φόρντ. Ευχαριστώ. Όταν ο Μπίσμπαρκ εισήγαγε το 1889 της Δημόσιας συντάξεις, το μέσο προσδόκιμο ηλικίας ήταν μόλις 45. Τώρα ζούμε περισσότερο, αντιμετωπίζουμε την πρόκληση. Πώ θα πετύχουμε να έχουμε επαρκή οικοδήματα κατά τη συνταξιοδότηση. Οι... Αλλάζουν πάρα πολύ οι παραδόσει οικονομικέ και κοινωνικέ. Επομένω, οι μεμονωμένε χώρε πρέπει να είναι υπεύθυνε για τι πολιτικέ του. Τα εφόρα κρατικά συνταξιοδοτικά συστήματα χρειάζονται επαρκή δημοσιονομικά, αλλά οι φάσει δεν μπορούμε να έχουμε εναρμόνιση του ορίου συνταξιοδότηση ή του ελάχιστου εισοδήματο τα εταιρικά σταξιδιωτικά συστήματα και τα ε, δυνατότητε επαγγελματικών ταμείων θα μπορούν να μεταφέρονται από το ένα εργοδότη στον άλλον και από μία χώρα στην άλλη. Θα πρέπει οι αποταμιευτέ να κατανορίζουν τι συνθήκε και να χρειαζόμαστε ασφαλή αποταμιευτικά συστήματα, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να είναι ευφυή κεφαλαιοποιητικά συστήματα. Γιατί βέβαια οι, οι αποταμιευτέ δεν μπορούν να έχουν όλη τη γνώση όπω οι τράπεζε, οι ασφαλιστικέ εταιρείε και επομένως δεν μπορεί η όλη προφόρηση να αντίχεται στον γυραίο, στον, στον πολίτη. Κυρία Σαρτιέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω πως η κρίση ε, και το πρόβλημα της δημογραφίας ε, αλληλεπηρεάζονται. Γιατί βέβαια ε, το πρόβλημα των συντάξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται πιο οξύ λόγω της κρίσης. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι γίνεται στην αγορά εργασίες, όπω επίσης και με το θέμα της διαβούλευση, το οποίο αναφέρθηκε ο επίτροπο κ. Όρμπαν. Θα πρέπει λοιπόν να διαβολευτούμε, να βρούμε μια δυνατότητα συμβιβασμού, ε, σύμφωνα με τα όσα είπε και η συγγήτρια, έτσι ώστε η ε, γνωμοδότηση αυτή να φτάσει ε, να ψηφιστεί. Υπάρχουν τρία σημεία τα οποία πρέπει να λάβουμε οπωσδήποτε υπόψη για να πετύχουμε ε, να εξασφαλίσουμε την φερεγγιότητα του συστήματος του συνταξιοδοτικού. Πρώτα απ' όλα η ανισότητα. Θύμα αυτής είναι σήμερα οι γυναίκες συνταξι... ηλικίες συνταξιοδότησης γιατί βεβαίως λόγω των περιορισμένων επαγγελματικών δυνατοτήτων και επαγγελματικής εξέλιξης ε, δεν έχουν τόσο ψηλούς μισθούς τη στιγμή που συνταξιοδούνται. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα γίνει με αυτή την γενιά των γυναικών που είναι φτωχές, για τις οποίες η βασική σύνταξη είναι ο μόνος τρόπος να έχουν μια ελά, ένα ελάχιστο εισόδημα. Έχουμε επίσης και τις νέες γενιές που αυτή τη στιγμή μπαίνουν στην αγορά εργασίας που έχουν να αντιμετωπίσουν όχι μόνο την κρίση αλλά και το βάρος των προηγούμενων γενναίων, αλλά και των μελλοντικών, δηλαδή των ε, ε, προγόνων τους, αλλά και των επιγόνων τους. Θα πρέπει λοιπόν να ε, δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε τα δικαιώματά τους χωρίς να μένουν για πάντα στην αγορά εργασίας. Η κυρία Στάινουρουκ έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι συντάξει θα πρέπει να υπαρκούν σε ολόκληρη την Ευρώπη και βεβαίω προπόθεση γι' αυτό είναι να υπάρχουν αξιοπρεπείς θέσει εργασία. γιατί οι φτηνέ δουλειέ οδηγούν σε φτώχεια και στην σύνταξη. Και αν κάποιοι εδώ πέρα θεωρούν πως ε, θα ασφαλιστούν οι άνθρωποι σε μια ιδιωτική σύνταξη πρέπει να σας ε, πληροφορήσω πως υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ζήσουν από τα λεφτά που βγάζουν πόσο μάλλον να πληρώσουν ιδιωτική ασφάλιση. Γι' αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία το αλληλέγγυο κρατικό συνταξιοδοτικό σύστημα και θα πρέπει να μπορεί να ζήσει κανείς από αυτό. Δεν μπορεί να λέμε πως είναι υπόθεση των κρατών μελών. Πρέπει να βγει από εδώ πέρα το μήνυμα πως χρειαζόμαστε συντάξεις με τις οποίες μπορούν να ζήσουν οι άνθρωποι. Ο συνάδελφος ο κύριος Τόμας Μάν αναφέρθηκε στο γερμανικό ε, σύστημα, ειδικά στην πτυχή της ε, επαγγελματικής σύνταξης. Κοιτάξτε, διαβάζοντας εγώ την ε, πράσινη βίβλο κατέληξα σε κάποια συμπεράσματα εξού και οι τροπολογίες οποίες ε, υποβάλαμε και θέλουμε άρα η Κομισιόν να λάβει υπόψη τις εθνικές ιδιαιτερότητες και αυτό είναι ζήτημα επιβίωσης για τα συνταξιοδοτικά συστήματα για να μην ξεμείνουν. Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κύριος Στολόγιαν για ένα μισή λεπτό. Ε, Uh, Νομίζω ότι πρέπει να φανούμε ρεαλιστές και να γνωρίσουμε ότι τα υφιστάμενα δημόσια εξωτερικά συστήματα που βασίζονται στην μεταφορά πόρων μεταξύ των γενεών, σύμφωνα με την αρχή της ε, σύνταξης σε διανεμητικό σύστημα, δεν είναι βιώσιμο σύστημα από οικονομική σκοπιάς. Από αυτή την έννοια λοιπόν τα συστήματα αυτά πρέπει να επιδοτηθούν από τους δημόσιους προπολογισμούς για να μπορούν να επιβιώσουν. Η γύρανση του πληθυσμού, η αυξημένη κινητικότητα των εργατικού δυναμικού επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τα ελλείμματα αυτών των δημόσιων αξιωτικών συστημάτων. Τα προτινόμενα μέτρα λοιπόν, είτε πρόκειται για παράταση του επίσημου ορίους ταξιοδότηση ή η αύξηση των ε, εισφορών, των κοινωνικών εισφορών, όλα αυτά τα μέτρα είναι περιορισμένη εμβέλεια. Και η κοινωνική αντίσταξη της αυτού του τύπου τα μέτρα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Νομίζω ότι είναι κατακλείδη πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η λύση είναι η μετάβαση του σταξιωτικού συστήματος στο οποίο ο ενεργός πληθυσμό κατά τη διάρκεια της ε, ε, ενεργού ηλικία τους θα δημιουργούν το δικό τους ε, συνταξιωτικό απόθεμα. Κύριος Κόζα, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευρωπαϊκή Ένωση απασχολείται με πάρα πολλά θέματα, με ανάπηρους κλπ. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για τα συνδεξιωτικά συστήματα, ακριβώς οι ανάπηροι είναι εκείνοι οι άνθρωποι που δεν καλύπτονται επαρκώς. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ε, Ε, δεν είναι κάτι το οποίο επέλεξαν να ενταχθούν στα συστήματα, τα συνταξιδοτικά της ε, αναπηρίας και βεβαίως ε, σε πολλές χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης τρέμουν τα θεμέλια του συνταξιοδοτικού συστήματος και βεβαίω αυτό είναι και αντίθετο με τη στρατηγική για την Ευρώπη 2020. Δεν μιλάμε ε, μιλάμε εκεί πέρα για την κάλυψη των αναγκών ε, των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ανάγκες ε, και δεν μπορούν να βρουν μια θέση εργασίας αυτοί οι άνθρωποι. Επίσης οι ευρωπαϊκές προβλέψεις δείχνουν πως θα πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή για το πως θα αντιμετωπίσουμε το ότι θα μειωθούν οι εργαζόμενοι και θα διπλασιαστούν ε, οι άνθρωποι οι οποίοι εισπράττουν εισφορές από το σύστημα. Ε, αυτό ειδικά αφορά και τους ανθρώπους με αναπηρία. Εγώ υποστηρίζω την ε, ιδέα της συγγήτριας που λέει πως έχουμε 50 εκατομμύρια ανθρώπους με ε, αναπηρία και 41% αυτών των ανθρώπων είναι εργαζόμενοι. Τι γίνεται με το υπόλοιπο 60%. Κάτι πρέπει να γίνει και με αυτού. Ευχαριστώ. Ο κύριο Ποπάκης για ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ την εισηγήτρια στην προσπάθειά τη να διατηρήσει τις απαραίτητες ισορροπίες μεταξύ τη οικονομική βιωσιμότητας και τη κοινωνική επάρκεια των συνταξιδοτικών συστημάτων όπου σε μια περίοδο υψηλή ανεργία, εργασιακή απορρίθμισης μισθολογικών περικοπών και έντονων δημογραφικών προκλήσεων η δημιουργία και εμπέδωση επαρκών κοινωνικά δίκαιων και οικονομικά βιώσιμων συνταξιοδοτικών συστημάτων αποτελεί μέγιστη πρόκληση για το κάθε κράτος μέλος. όμως ο πρώτος πυλώνας ο δημόσιος αναδιανεμητικός χαρακτήρας οφείλει να είναι το επίκεντρο των συστημάτων μοναδικός βασικός εγγυητής τη επάρκεια των παροχών και, όχι συνεπικορούμενο από το δεύτερο πυλώνα που θα πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά αφού προηγούμενα διασφαλιστεί όχι μόνο η πρόσβαση όλων σε αυτόν αλλά και η ασφάλειά του με καθιέρωση σχετικού πλαισίου διακυβέρνηση. πέρα από αυτό διασύνδεση επέκταση εργασιακού βίου και προσδόκιμου ζωή δεν μπορεί επουδενή να οδηγεί σε αυτόματε προσαρμογέ. σε κάθε περίπτωση βέβαια θα πρέπει να συνυπολογίζονται και άλλοι παράμετροι όπω γεωγραφικά χαρακτηριστικά φύση τη εργασία βαρέα ανθιγεινά επαγγέλματα ποιότητα ζωή και υγεία. ενώ τέλο τα όποια κίνητρα παραμονή στην εργασία θα πρέπει σαν προϋπόθεση να εμπεριέχουν τέτοιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να μην παροκολύουν την πρόσβαση των νέων στην αγορά εργασίας σε μια περίοδο μάλιστα που η ανεργία φτάνει δυστυχώς σε δυσταιόρατα ύψη. ευχαριστώ. κύριε και ξεκινάει η συζήτηση Catch the Eye, αλλά οφείλω να σας πω ότι έχουμε αρκετή καθυστέρηση γιατί συντομεύσαμε κατά μισή ώρα τις ερωτήσεις προς την Επιτροπή λόγω των άλλων θεμάτων που παρευλήθησαν. Έχω 17 αγορητές του λόγο. Μόνο 5 θα πάρω για να κρατήσουμε και κάποιο χρόνο συζήτηση για την επόμενη έκθεση για τα παραπημένα φάρμακα. Θα προσπαθήσω να κρατήσω κάποια ισορροπία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων και ξεκινώ δίνοντας το λόγο στον κύριο Ρούμπικ από το ΕΛΚ. Έφυγε, καλό ή κακό για τον ίδιο. Με δεδομένο ότι δεν είναι εδώ λοιπόν. Η κυρία Λουκασιζέφικα. Przewodnicząca, dyskusje, jak odbywają się w niektórych krajach Unii Europejskiej na temat systemów emerytalnych. I όλη η συζήτηση που είναι σε εξέλιξη στις, ε, στα κράτη-μέλη σχέση με τις συντάξει και με τις μεγάλες κοινωνικές πιέσεις ε, οι μεγάλε πιέσει που υπάρχουν καταδεικνύουν πόσο δύσκολο είναι το θέμα. Δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ένα ενιαίο μοντέλο συντάξεων που θα μπορεί να είναι υποχρεωτικό σε όλε τι χώρε. Όμω, με δεδομένη ε, τη ε, μεγάλη δημογραφική κρίση, η μεταρρύθμιση των εθνικών συνταξιδοτικών συστημάτων είναι αναπόφευκτη. Πολλέ χώρε αντιμετωπίζουν προβλήματα με τον αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων και βέβαια αυτό μπορεί να διακυβεύει το όλο ζήτημα ε, αλληλεγγύη όμως οι συντάξεις θα πρέπει να είναι εξασφαλισμένες λαμβάνοντα υπόψη τις ε, απολαυέ μα, του επίπεδου των ε, μισθών μας. Επισημαίνω λοιπόν και πιστώ την προσοχή σα στι ανισότητε που υπάρχουν μεταξύ γυναικών και ανδρών, γιατί η χαμηλή μισοδοσία των γυναικών προφέρει και πολύ χαμηλέ συντάξει. Ευχαριστούμε. Η κυρία Πλούμπ για ένα λεπτό. Είναι εδώ. Έχει το λόγο. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να πω ότι ακόμα και στην αρχή της συζήτησης ο εισηγητής μιλούσε για την επιτυχία του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου και μία, ένα από τα συνιστόντα στοιχεία αυτής της επιτυχίας είναι ακριβώς η ισότητα ευκαιριών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Ελπίζω λοιπόν ότι η έκθεση αυτή θα μπορεί να μεταφέρει ένα σαφές μήνυμα σε ό,τι αφορά την ένταξη της συνιστώσεως αυτής, ε, της ισότητας ευκαιριών σε ένα σωστό σύστημα συνταξιοδότησης. Και τονίζω τρία σημεία. Θέλω να μιλήσω για την ανάγκη αποτίμησης του αντίκτυπου που έχει στην κοινωνία τα διάφορα μέτρα αναγνώρισης της κατοίκων εργασίας λαμβάνοντας ακριβώς υπόψη έναν χρηματοοικονομικό υπολογισμό για να αποτιμηθεί αυτή η εργασία, η κατοίκον εργασία, η προσφορά ε, στο σπίτι στην σχηνική σύνταξη. Και αυτό ζητώ από την Επιτροπή να καταργήσει την ε, παραγράφο 5 ε, στην οδηγία που θέτει το ζήτημα συντάξεως των γυναικών. Το Ευχαριστώ πολύ. Το συνταξιδοτικό σύστημα στην Ευρώπη είναι ένα από τα βασικά κοινωνικά κεκτημένα της Ευρώπης για να επιβιώσει. Πρέπει να λάβουμε μέτρα με τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας και των κοινωνικών εταίρων, ώστε να έχουμε ένα πρότυπο ευρωπαϊκό που θα εξασφαλίσει τη φερεγκιότητα όλων των συστημάτων, βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη εποπτείας των δημοσιονομικών συστημάτων στην Ευρώπη και βεβαίως θέτοντας κάποιες επι απαιτήσει από το 2013 στις ασφαλιστικές εταιρείες και στα ιδιωτικά ταμεία που υπάρχουν σε κάποια κράτη-μέλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο και να κάνουμε κάτι παραπάνω από το απλώς να ορίσουμε ε, το όριο της ηλικίας συνταξιοδότησης. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε και ποιους άλλους παράγοντες θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη, παράδειγμα προωθώντας, δίνοντας κάποια προνόμια στους εργαζόμενους οι οποίοι παραμένουν στην αγορά εργασίας μετά την ηλικία συνταξιοδότηση. Να δούμε τι γίνεται με τη μεταφορά συντάξεων από χώρα σε χώρα. Και θα πρέπει να μπορεί ένα εργαζόμενο να λάβει στη σύνταξή του όλε τι εισφορέ που έχει πληρώσει όπου και αν δουλεύει στην Ευρώπη. Η κυρία Στρούντερ έχει το λόγο μετά την κυρία Μπιλμπάου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Αναρωτιέμαι εάν πραγματικά έχει νόημα να απαντήσουμε πάλι με μια λευκή βίβλο σε αυτή τη συζήτηση και να μην λύσουμε τα κατεπήγοντα προβλήματα, τα οποία είναι δύο. Πρώτον, βλέπετε πως η πραγματική και η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης διαφέρουν κατά πολύ. Πρέπει επίσης να υπάρξει καταπολέμηση των διακρίσεων από την Κομισιόν με ελέγχου της Κομισιόν για να βελτιωθεί η κατάσταση, για να είναι βιώσιμες συντάξεις και δεύτερον ζητήστε κάντε κάτι ειδικά όσον αφορά το να μπορούν να μεταφέρονται διασυνοριακά οι συντάξεις με την οδηγία την οποία φέρνετε τώρα. Αυτό είναι κατεπήγον γιατί υπάρχουν μετακινούμενοι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν λεφτά από τη σύνταξή τους για μια πιο σίγουρη ζωή. Και χάνουμε πάρα πολύ χρόνο εδώ πέρα άμα ασχολούμαστε με λευκές βιβλίες. Ευχαριστώ κύριος Ρούμπιξ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, σε καιρούς ε, οικονομικής ε, κρίσης, ως ε, αποτέλεσμα της διαδικασίας γύρανσης βλέπετε πως οι κοινωνικές παροχές μειώνονται, ο αριθμός των συνταξιούχων αυξάνεται και αυτό βεβαίως υπονομεύει την βιωσιμότητα του συστήματος σύνταξης, οπότε θα πρέπει να το προσαρμόσουμε στις ε, τωρινές ε, προκλήσεις και συμφωνώ με τον Επίτροπο που είπε πως θα πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να αναπτύξουμε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές. Θεωρώ όμως πως θα πρέπει να υπάρξει ένα κοινωνικό ταμείο παρόμοιο με το Ταμείο Συνοχής για να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν χαμηλό εισόδημα και εκεί όπου ο κρατικός περιπολογισμός δεν μπορεί να διασφαλίσει επαρκές εισόδημα για τους ηλικιωμένου. Και βλέπετε πως αυτοί είναι όλο και περισσότεροι. Ζητώ συγγνώμη από τους υπόλοιπους για τον λόγο, αλλά πρέπει να δώσουμε το λόγο στον ε, Επιτροπό, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ακούσουμε τι έχει να μας πει σε όλες αυτές τις αιτιάσεις. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε πολύ. Θέλω Θέλω να συγχαρώ και πάλι τις επιτροπές, όλους όσους συμμετέσχουν στην όλη συζήτηση και στην, σε όσους λύσαν την εισήγηση, καθόλου και την εισηγήτρια. Δεν είναι δυνατόν να απαντήσω στις θέσεις, ε, βέβαια, και να ευθυγραμμιστούν όλες αυτές οι διαφορετικές θέσεις ε, από διαφορετικά κράτη-μέλη. Αλλά βλέπουμε ότι οι ψηφοφορίες που δοθούν μας στέλνουν σαφή μηνύματα για την παρακολούθηση της πράσινης βίβλου. Ε, αρχές του επόμενου μήνα θα δοθεί μια σύνοψη περιλαμβάνοντας και τις συμπεριλαμβάνοντας τροπολογίες από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στο δεύτερο εξάμεινο του 2011 θα δημοσιευθεί η λευκή βίβλος στην οποία ανέφερα στην αρχή που θα συνοδεύεται με μια αντίστοιχη ε, ε, έκθεση αξιολόγησης των επιπτώσεων. Αυτό θα οδηγήσει όλους τους εμπλεκόμενους να συνεχίσουν να μετέχουν ενεργά στην όλη συζήτηση. Μπορώ να σας προφορήσω από τώρα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα εξωτικά ζητήματα ήδη συζήτησε το πώς μπορεί να ενημερωθεί και να επικαιροποιηθεί το υφιστάμενο πλαίσιο. Υπήρξε συμφωνία να συνεχίσουμε στο φόρουμ αυτό με την ολιστική προσέγγιση σε ό,τι αφορά τη μεταρρύθμιση εξωτικών συστημάτων. Πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με τους κοινωνικού εταίρους και για ενδυνάμει νέε νομοθετικές ε, προτάσεις σε ό,τι αφορά την μεταφορά δικαιωμάτων και παροχών και προστασία μέσω της φερεγγιότητας και άλλες μορφές ε, ε, νομοθεσίας, κανονισμού, όπως είναι με αυτό με τις καλές πρακτικές. Επίσης συζητήσαμε εις βάθος και θα συνεχίσουμε να συζητούμε τα θέματα ε, ανισοτήτων μεταξύ των φύλων και θα συμπεριληφθούν και στη Λευκή Βίβλο. Εν τω μεταξύ, θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι και η Πράσινη και η Λευκή Βίβλο δεν θα πρέπει να, δεν θα πρέπει να μπερδεύονται μεταξύ τους, αν θέλετε, σαν κάτι τελείως άστο μεταξύ τους. Θα πρέπει να υπάρχει μια ενιαία... Ε, δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ενιαίο ηλικία ταξιοδότηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ποικιλία είναι βασική στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ισχύει και στη δημογραφικά. Και πρέπει να μελετήσουμε πολύ πιο βαθιά το θέμα αυτό από ό,τι στο παρελθόν. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι ενεξελίξεις μετερρυθμίσεις φέρουν περισσότερους κινδύνους, γιατί κάνουν ακόμα πιο τα στοιχεία και παράγοντες με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και στα δημογραφικά. Πρέπει να δημιουργηθούν ευκαιρίες απασχόλησης και για τα άτομα με ειδικέ ανάγκες και να αυξηθεί η σταθερότητα των χρηματοοικονομικών συστημάτων. Αξιότιμο μέλη, θα, Προσβλέπω τη συνέχιση συνεργασία μαζί σα, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή και τι αρμόδιε επιτροπέ, πάνω στο πολύ σημαντικό αυτό ζήτημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και ολοκληρώνουμε συζήτηση με την εισηγήτρια, την κυρία Όμεν Γόιτα. Δράτω τη ευκαιρία για να κατονομάσω τους συναδέλφους Γκέρ Κούτας, Μπάρμπαρα Ματέρα και τον κύριο Ντε οι οποίοι έκαναν κάποιες παρατηρήσεις τις οποίες ε, δεν ε, αντιλαμβάνομαι πλήρως. Ε, ε, λέτε ότι θέλω να τα λύσω όλα ευρωπαϊκά. Όχι. Η αρχή είναι η επικουρικότητα. Κύριε Πρόεδρε, το πρόβλημα τώρα που υπάρχει με την οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι ο καθένας να κάνει ό,τι μπορεί για να έχουμε θετικά αποτελέσματα στην οικονομική διακυβέρνηση. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε κάποια κράτη-μέλη τα οποία έγραψαν αυτή την επιστολή να βρεθούν σε δυσμενέστερη θέση γιατί φροντίζουν για ένα καλό μέλλον, για τις ε, συντάξεις. Η κυρία Λιωτάρ δεν είναι εδώ πέρα, αλλά αντιλαμβάνομαι πως προφανώς δεν διάβασε την έκθεση αλλά εξακολουθεί να κάνει δηλώσεις χωρίς κανένα πρόβλημα. Ανέφερα ήδη τους ε, τρεις ε, συναδέλφους, οποίους ευχαριστώ, αλλά να αναφέρω και του Τζουλ Γκέρλινγκ, Τζιν Λάμπερτ, την Ντανούτα, την δική μας ε, σκιώδη για το ότι με βοήθησαν σε αυτή την έκθεση για να γίνει αυτό το οποίο είναι. Επίσης, νομίζω ε, πως έγιναν καλές αναλύσεις για το τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και μπρος. Ξέρω πως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ευαισθησίες που σχετίζονται με τα κράτη-μέλη, αλλά παρόλα αυτά θεωρώ πως ε, είναι καλό το έργο το οποίο κάνετε εδώ πέρα, κύριε Άντερ, και νομίζω πως θα πρέπει να προχωρήσουμε στη Λευκή Βίβλο για να ακολουθούμε όλοι μία κοινή γραμμή σε αυτό το κοινοβούλιο. Ήταν δύσκολη αυτή η υπόθεση. Ελπίζω λοιπόν αύριο να μπορέσουμε να την υπερψηφίσουμε και να πούμε τέλος καλό. Όλα καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κυρία Όμεν Και εδώ πέρα τελειώνει η συζήτησή μας. Ψηφοφορία αύριο το μεσημέρι. Για όσους δεν μίλησαν, εάν το επιθυμούν, μπορούν να υποβάλουν μια γραπτή εξήγηση η οποία θα